Président. Mesdames, Messieurs, Madame la Commissaire. Κυρίες και κύριοι, κυρία Επίτροπε, επαναλαμβάνεται η σύνοδός μας. Αρχίζω με τα πρακτικά, τα χθεσινά πρακτικά, για να σας πω ότι είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Φαίνεται πως όχι, άρα τα πρακτικά εγκρίνονται. Επίσης έχω μία ανακοίνωση από